Ο Πρόεδρος. Άρχεται η συνεδρίαση. Το πρώτο θέμα της ημέρας της διάταξης είναι η δήλωση Συμβουλίου και τη Επιτροπή για την προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου